έργο. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει αύριο, Τρίτη, σε 9 το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ.